Allora iniziamo. Chiediamo scusa per qualche minuto di ritardo causa un rischio Παραλίγο να ανατραπούν όλα. Να δυναμιστεί η συνάντησή μα γιατί παραλίγο να μα πάρουν του τερμίδε να πάνε κάπου αλλού. Όμω δεν έγινε αυτό και έτσι ευτυχώ τώρα αρχίζει η δουλειά μεγάλη με ευχαρίστηση, Καλώ όρισαν οι Ούγγροι προσκεκλημένοι μας. Του εύχομαι καλή διαμονή. Και ιδίως αμέσω να προβούμε στην έγκριση των πρακτικών της Για να δεν έχετε παρατηρήσεις ενστάσεις, τότε να θεωρηθούν εγκεκριμένα. Και εάν δεν υπάρχει κάποια ένσταση θα είναι οριστικά εγκεκριμένα τα πρακτικά της συνεδρίασης και ε, μεταδίδεται στην συνεδρίαση μέσω του web stream. Ευθύς αμέσως προχωρούμε εις την ψηφοφορία. Πολιτική βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την παραγωγή βοήθεια από τι όμορφε χώρε προ αντιμετώπιση προκλήσει τη επισητιστική ασφάλεια. Μάρκ Ταραμπέλα είναι ο εισηγητή. Και ευθύ αμέσω προχωρούμε στην ψηφοφορία. Μάρκ, θέλεις το λόγο. Μιλάω να πάμε να ψηφίσουμε. Ταραμπέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μπορούσα να πω πολλά αλλά θα περιοριστώ να χαιρετήσω όσους συνεργάστηκαν εδώ και δισκιώδης ιδίω γιατί πετύχαμε έξι συμβιβασμούς σίγουρους και υπάρχουν και άλλες τροπολογίες βέβαια. Χαιρετίζω επίσης όλους όσους συνεισέφεραν στην εργασία αυτή, όχι μόνο συναδέλφους, αλλά και τους υπαλλήλους, Σόνια Στέλλο, τη Μαρία Πάολα, Ντιάντζελη, Σόρενσεν, Γκούναουτσου και άλλους, που δεν τους αναφέρουμε συνήθως ποτέ, αλλά δουλεύουν στη σκιά. Επίσης, ο κατάλογος της ψηφοφορίας είναι πολύπλοκος γιατί πρέπει να γνωμοδοτήσουμε προς την Επιτροπή Ανάπτυξης γιατί θέλαμε να επιμείνουμε θα τα πει και ο συνάδελφος Σιλβέστρης, ίσως να τα πει και πιο στεναρά και από μένα για τα διαδικαστικά, για το χρονοδιάγραμμα κάποτε έπρεπε να σταματήσουμε και αυτό θα το ξαναδούμε επειδή υπάρχουν συμβιβασμοί που δίνουν ένα ασχελτρά αρκετά ισχυρό μήνυμα. Θα ήθελα να φέρω ιδιαίτερα την κυρία Πατράου Νέβες που ευχαριστώ, την κυρία Νταντσίλα από την ομάδα μου και άμα βλέπετε μείον σημαίνει ότι είμαι κατά. Αλλά πολλές φορές δεν είμαι βέβαιος. Απλώς προσπάθησα να τα πω καθαρά και προσωπικά μπορώ να δεχτώ ορισμένες ιδέες αλλά δεν θέλω να διαλυθεί, να αραιωθεί το κρασί μας με αυτές. Γι' αυτό τις έχω ζητήσει να καταψηφιστούν. Δεν είναι αποχρεωτικά ότι διαφωνώ. Καταψηφίζω μερικές τροπολογίες αλλά σε πνεύμα έτσι για να μείνει συνοπτική η έκθεση και να μην αποδυναμωθεί. Γι' αυτό μερικές τροπολογίε τις έχω βάλει μείον. επαναλαμβάνω ότι ευχαριστώ όλου του συναδέλφου που έχουν συνεισφέρει σε αυτή την εργασία διότι για μια τέτοια γνωμοδότηση χρειάστηκαν πολλές ανταλλαγέ απόψεων και α σταματήσω εδώ για να μην μακρο, μακρηγορήσω τυχόν. ευχαριστούμε λίγο Πρόεδρος και ευθύ αμέσω ταχαίως προχωρούμε στην ψηφοφορία. Αρχίζουμε. Έχετε όλη την λίστα. Όχι. Και την, κάρτα. Όχι. Δεν έχει την ηλεκτρονική κάρτα ο Κάπουλα Σάντο. Να σημειωθεί αυτό και, πάμε, και ξεκινούμε την πρώτη τροπολογία. Ε, Χωστή ψηφορία σε τρία κομμάτια. Πρώτο κομμάτι Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για το δεύτερο τμήμα της πρώτης τροπολογίας. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Τέλος. Το τρίτο τμήμα. Πέρας. Απορρίπτω. Πολύ ωραία. Δεύτερη τροπολογία. Σιλβέστρης. Ψηφίζουμε. Πέρας. εγκλίνεται. Τρίτη. Σε δύο τμήματα. Το πρώτο. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, τροπολογία 3. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Πάμε στο 6. Ψηφίζουμε. Τροπολογία 6. Πέρας. Απορρίπτεται. Ah allora, chiedo scusa, votiamo il συμπαθάτε με. Θα ψηφίσουμε τώρα το 5 το οποίο το παραλείψαμε. Ψηφίζουμε το 5. Πέρας Εκεί, εγκρίνεται. Επόμενο εντάξει είναι το 5 και το 6 το κάναμε. Πάμε στο 7. Ψηφίζουμε το 7. <coughs> Edward. Chiusa la votazione sul 7. Πέρας. Απορρίπτεται. 8. Πέρας ψηφοφορίας για το 8 και εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε παριθμό 10. Για 10. Ψηφίζουμε. Πέρας. Αδοτάτο. Εμενταμέντο. Εγκρίνεται. 11. 11. Πέρας. και εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε όλα τα σχετικά με την συμβαστική 1. Πέρας. Εγκρίνεται η συμβαστική παριθμόν 1. 19. Πάμε στην 19. Πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19, δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας και εγκρίνεται. Η 21 πατράων 21 ψηφίζουμε. Πέρας. 21 εγκρίνεται. 22 ψηφίζουμε. 22 πέρασε. Α, απορρίπτεται. Τροπολογία 24 εις 2 τμήματα το πρώτο. Ψηφίζουμε. Πέρας. Έγκρινεται. Και τώρα το δεύτερο τμήμα. Το 24. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 25. Πέρας. Απορρίπτεται. 26. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 27. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. 28. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 29. Πέρας. Εγκρίνεται το 29. Και τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 30. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την συμβαστική υπαριθμών 2. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στο 36. Λάιον και άλλων. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε το 39. Το 39, ψηφίσουμε το 39. Πέρασε. Α, απορρίπτεται. 45. Ψηφίζουμε. Πέρας, απορρίπτεται. Είπαμε τώρα στην συμβαστική 3. Εις δύο τμήματα. Πρώτον, ψηφίζουμε. Πέρας. Το πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής 3. Πέρας. Εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία περιθμών 55. 55. Νικουλέσκου. Πέρας. Σας πέμψ. Αγωνία λέει πρόεδρος και απορρίπτεται. Noi ti abbiamo sostenuto. Andiamo al compromesso 4. parametro τώρα στην συμβαστική 4. Ψηφίζουμε. Θέλετε το, το λόγο κύριε Σιλβέστρη. Εκτό μικροφώνου κύριε Σιλβέστρη. Δεν ακούγεται τι λέει. Θα σα την παρουσιάσω μετά την ψηφορία. Ναι, ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε τη συμβαστική Τέσσερα. Ψηφίζουμε. Σε la votazione sul 4. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον ε, κύριο Συντλέστας για μια προφορική τροπολογία την οποία και θα μα κατεβάσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγγνώμη που να βάλω τον ε, λόγο γιατί πρόκειται για αυτή την προφορική τροφολογία αλλά ε, μου έχουν πει ότι πρέπει να επιμείνω γιατί πρόκειται μια προφορική τροπολογία την οποία και σας προτείνω και θα αντικαταστεί στο δεύτερο τμήμα τη συμβαστική τροπολογία που τώρα εψηφίσαμε με ένα κείμενο το οποίο νομίζω ότι το έχετε λάβει. Και δεν ξέρω εάν ε, έχετε μπορέσει να το διαβάσετε και τι θέλω να πω. Θέλω να συνδέσω κάπως ούτω ώστε να συνδέσουμε αυτό το πρόγραμμα βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και αυτό να μας βοηθήσει στην γεωρική παραγωγή και έτσι ε, από πλευρά ενεργειακής να υπάρχει αυτενέργεια και να έχουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα ούτω ώστε να έχουμε κάποιες ανεώσιμες ποιε ενέργειας οι οποίες εκεί να πιάσουν τόπο και έχουμε κάποιες καθολικέ οργανώσεις, ε, κάποιε αποστολέ, ιεραποστολέ και όλοι αυτοί προσπαθούν εκεί να βοηθήσουν σε διάφορες μειονεκτούσες ε, περιοχές της Υπέθρου. Όταν όμως ε, έρχεται η, η ώρα της χρηματοδότησης, οι εγκαταστάσεις που εκεί έχουν δημιουργηθεί εγκαταλείπονται. Άρα, να μην χρηματοδοτήσουμε μόνο την καλλιέργεια κάποιων προϊόντων, κάποιων φυτών, αλλά να υπάρχει χρηματοδότηση για τις ε, κατάλληλες εγκαταστάσεις, ούτω ώστε να μπορέσουμε να οδηγήσουμε αυτές τις χώρες προς την αυτάρκεια. Ευχαριστώ. Και τώρα ζητεί τον λόγο ο εισηγητής ο κύριος Ταραμπέλα. Έχεις τον λόγο. Πρόεδρε, ήθελα να πω ότι το πρόβλημα με αυτή την τροπολογία δεν είναι το περιεχόμενο, γιατί υπερβαίνουμε ε, ουσιαστικά αυτό που είχαμε επιδιώξει αρχικά. Οπότε, επί της ουσίας, ε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά με τον κύριο Σιλβέστρη και τον κύριο Έλκορντ, Όσλινγκ, Φοντάνα και Άσφορντ, ε, είχαμε συμφωνήσει για τον τύπο της τροπολογίας 4. Δηλαδή, σήμερα στο 12.30 δεχτήκαμε αυτή την προφορική τροπολογία και δεν ήρθα σε επαφή με τις λοιπές πολιτικές ομάδες για να αλλάξουμε τα πράγματα τελευταία στιγμή. Αυτή η συμβαστική ε, τροπολογία ε, έτυχε ούτως άλλως αποδοχής ε, όλων των πολιτικών ομάδων. Είναι τυπικό το θέμα, δεν είναι ουσιαστικό. Για τη διαδικασία πάντως θα πρέπει να μεριμνήσουμε τόσο ώστε να μην επαναληφθεί αυτό, γιατί στις 2 η ώρα συνεδρίασε η ομάδα εργασίας. Η προβλήμα, Μάρκ. Μάρκ, λέει ο πρόεδρο, άκουσε με. Το πρόγραμμα είναι ότι εάν εσύ θέλει ψηφίσουμε. Γιατί αν είσαι ενάντια, ξέρω με τον κανονισμό, δεν θα γίνει η ψήφιση. Ε, για να είμαστε σωστοί, επειδή εργάστηκαν όλοι, να ψηφίσουμε αυτή την τροπολογία. Ούτω ή άλλω, επί του περιεχομένου συμφωνώ. Ήθελα να κάνω μόνο αυτή την παρατήρηση επί τη διαδικασία. Δεν μπορούμε να εργαζόμαστε έτσι. Σέβομαι όλου όσου εργάστηκαν ε, και τα, τη λάβαμε δύο ώρε πριν από την ψηφοφορία. Ε, συμφωνώ, εν πάση να ψηφίσουμε για αυτή την τροπολογία. Άρα, τώρα θα ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία όπω μα την εξέθεσε ο κύριος Σιλβέστρη. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό που ο κ. Ταραμπέλα, ψηφίζουμε τώρα την προφορική τροπολογία. Bene, dichiaro chiusa Πέρας. προφορική τροφολογία και τώρα. 61, Πατράο Νεβές. 61 ψηφίζουμε. Το 61. Sulla votazione sul 61. 61. Εγκρίνεται. Το πρώτο τμήμα του 62. Ψηφίζουμε. Πρώτο τμήμα. 62. Πέρασε. Πέρας. Απορρίπτεται. 64. Τώρα το 64. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα πάμε στην συμβαστική 5. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Εβδομήντα επτά. Λέω πρώτος και τώρα το πρόθυμα του εβδομήντα επτά. Δεύτερο τμήμα τώρα του 77. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα του 77. Πέρας. Εγκρίνεται. Chiusa la votazione sul 78. Adottato. Εγκρίνεται το 78 και πάμε στο 79. Πέρας. Εγκρίνεται. 80. Πέρας. Εγκρίνεται. 81. Γκλάτφελντερ. Ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Σιλβέστρης για να παρουσιάσει την προφορική τροπολογία σε σχέση με το 82. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν είναι κείμενο που δεν το έχουμε εδώ, γιατί θέλουμε εδώ ή στην παράγραφο 8 να πούμε ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις τοπικές αρχές να μπορούν να διεξάγουν διαπραγματεύσεις όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου κλπ. κλπ ούτως ώστε να είναι δυνατόν κάποιες επενδύσεις για εγκαταστάσεις που αφορούν τη γεωργία που θα βοηθήσει να ζει καλύτερα ο πληθυσμός υπαίθρου. Τα είπατε πάρα πολύ γρήγορα και δεν μεταφράστηκαν. Εύκολα. Και τώρα. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε όσον αφορά αυτήν την τροπολογία. Όπως μόλις μας την εξήγησε ο συνάδελφος, ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι ε, για το 82. Εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε την 83. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεύτερο τμήμα της συμβαστικής 6. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα συνεχίζουμε με το 63. Ψηφίζουμε. Πέρας. Ο 84. Πέρας. Εγκρίνεται. 85 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα του 85. Πατράω νεύες. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Azione. Respinto. Πέρασε. Και απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα του 85. Ε? ε, και το σκούσα. Ακόλτο. Ακόλτο. Α, όχι. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Συμπαθάτε με το πρώτο. Το πρώτο τμήμα του 85 εγκρίνεται, διορθώνει ο πρόεδρο. Και τώρα το δεύτερο τμήμα του 85. Ε, Credo la stessa maggioranza. Νομίζω ότι συνεκέντρωσε την ίδια πλειοψηφία και επομένω και αυτό το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται και τώρα. Μισό λεπτό. Πάμε στο 87. Ψηφίζουμε το 87. Πέρας. Και αυτό μου φαίνεται όμως ότι απορρίπτονται. Και πάμε στο 88. Μάλλον εγκρίνεται. 89. Εγκρίνεται και αυτή η διάταξη. Και ψηφίζουμε τώρα το 90. Μάνερ. Ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. 91. Πατράων Εύες. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. 54. Ψηφίζουν το 54. Πέρας. Εγκρίνονται. 92. Πρώτο τμήμα. Πέρας. Το πρώτο τμήμα απορρίπτεται. Και τώρα το δεύτερο. Το 92. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στο 93. Ψηφίζουμε. 93. 93. Πέρας, απορρίπτωται. Τώρα έχουμε την καταληκτική ψηφοφορία και επομένω ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου ω τροποποιήθηκε. Πέρα. Έγκρινεται ναι. συγχαρητήρια ει τον κύριο Ταραμπέλα. Ευχαριστούμε συνεργατικά και στον κύριο όμως. Και πάμε τώρα, μιλήσω στο σημείο 5 της μέσας και το οποίο αφορά την έλλειψη πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η λύση για ένα τέτοιο μακροχρόνιο πρόβλημα. Ο εισηγητής είναι ο Μάρτιν Χόισλινγκ, είναι ένας βασικός στόχος του κειμένου του κυρίου Χόισλινγκ είναι το να αναδείξει το πόσο χρειάζεται να ληφθούν κάποια μέτρα και μέσα πολιτικής ούτως ώστε να βοηθήσουμε την παραγωγή πρωτεϊνών σε σχέση με τα νομοθετικά μέτρα που έχουν ε, σχέση με τη σειρά με την μεταρρύθμιση της Κάπκυρε Χόισλινγκ για το λόγο. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλους. Ο, για όσους έμειναν μέσα στην αίθουσα μετά την ε, ψηφοφορία, Ε, το θέμα αυτό εγγράφεται στα πλαίσια της νέας ε, κοινή γεωργικής πολιτικής και είναι ένα πρόβλημα που χρονίζει και οξύνθηκε, ε, μάλλον παρά το πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Ε, έχουν εγκαταλειφθεί οι πρωτεϊνικές ε, καλλιέργειες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο 3% της αρωτρέας γης καλύπτεται από πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και σε χώρες όπως η Γερμανία η έκταση που καλύπτεται ανέρχεται μόνο στο 1%. Ε, οπότε χρησιμοποιούνται πολλές φυτικές πρωτεΐνες. Ε, περίπου 80% των εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπετε λοιπόν σε ποιο σημείο εξαρτώμεθα από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Ε, κινητοποιούμε 20 εκατομμύρια εκτάρια για την καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνολική μας παραγωγή σχεδόν εξαρτάται από αυτή την εισαγωγή των πρωτεϊνούχων και άρα βρισκόμαστε σε μια επισφαλή θέση. Δεν είμαστε οι μόνοι βέβαια που ε, το κάνουμε αυτό και η Κίνα ε, ε, εισάγει εξίσου. Βλέπετε λοιπόν ότι διατρέχουμε ένα κίνδυνο αποσταθεροποίησης. Φυσικά υπάρχουν και ιστορικοί λόγοι που αιτιολογούν την ύπαρξη αυτού του πρωτεϊνικού ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα η Συμφωνία Γκάτε, η Συμφωνία Blair House, οδήγησαν σε αυτό το έλλειμμα γιατί επηρεάζουν τον ανεφοδιασμό μας σε ε, πρωτεΐνες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παραγωγή σιτηρών τελικά επηρέασε αρνητικά την παραγωγή πρωτεϊνούχων. Ε, έχουμε λοιπόν ουσιαστικό πρόβλημα, μπορεί να αναρωτηθεί κανείς. Βεβαίως, ε, ε, μακροπρόθεσμα θα χάσουμε τις παραδοσιακές πρακτικές καλλιέργειας των πρωτεϊνούχων και τα όσπρια καλλιεργούνται πολύ λιγότερα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάνουμε λοιπόν αυτή την τεχνογνωσία στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε αυτά τα φυτά για την ε, κτηνοτροφία, για, την, ε, για τα φυτόρια, για, τις, για, τις, ε, για την παραγωγή σπόρων, είναι καταπήγον το ζήτημα, πρέπει οπωσδήποτε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο αν δεν θέλουμε να τα χάσουμε όλα. Η βιομηχανία σπόρων επίσης εξαρτάται από αυτό και άρα πρέπει να θέσουμε πάλι σε λειτουργία το μηχανισμό και να αναπτύξουμε και νέες ποικιλίε ε, βελτιωμένες φυτικές ε, ποικιλίε. Ε, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης κοινή γεωρικής πολιτικής, ε, ποια είναι η βαρύτητα των πρωτεϊνικών καλλιεργειών. Ε, σας είπα ότι το παρόν ζήτημα εγγράφεται πλήρως στα πλαίσια των στόχων της νέας κοινής γεωρικής πολιτικής διότι αυτές οι καλλιέργειες είναι πολύ πιο οικολογικές, πολύ πιο βιώσιμες. Οι πρωτενιούχοι σπόροι, τα όσπρια δεσμεύουν 300 κιλά αζότου αναζώνη ανά εκτάριο ε, και έτσι ε, δεν ε, ε, εξαπλώνονται τα αζωτούχα λιπάσματα και επίσης υπάρχει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Θα πρέπει όλα αυτά να συνυπολογιστούν όταν θα συζητήσουμε το μέλλον της κοινή γεωρικής πολιτικής. Για όλους αυτούς τους λόγους βλέπετε πόσο κρίσιμο είναι το ζήτημα για το μέλλον. Δεν μιλάμε μόνο για την επάρκεια, την επισητιστική επάρκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μέλλον, όταν θα έχουμε αναθεωρήσει την κοινή γεωρική πολιτική, πρέπει να επωφεληθούμε από τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν αυτές οι καλλιέργειες ε, για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των καλλιεργειών και για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Ε, για την ε, πρωτεϊνούχο χορτονομή υπάρχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Νομίζω ότι για την βιομηχανία θα πρέπει να διευρύνουμε τις δυνατότητες αποθήκευσης ε, των ζωοτροφών. Επίσης, ε, να έχουμε τη δυνατότητα χρήσης ε, μειγμάτων ζωοτροφών και να προσανατολιστούμε επί τη βάση αυτών των στοιχείων για να καταρτήσουμε τη μελλοντική μας πολιτική. Μην ξεχνάτε επίσης και τις καλλιέργειες σόγιας. Δεν είναι αμελητές σε πολλές χώρες, όπως στην Αυστρία παραδείγματο χάρη. Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε σημαντικά η καλλιέργεια της σόγιας. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα διατηρηθεί ε, αυτή η τάση στο μέλλον. Η Γαλλία και άλλες χώρες προσπαθούν να ενθαρρύνουν την άσκηση της των καλλιεργειών αυτών και μπορούμε να δούμε ε, ε, πώς ενδεχομένως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη θετική γαλλική εμπειρία και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνω επίσης να θεωρεί να γίνουν υποχρεωτικές αυτές οι καλλιέργειες εφόσον χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζωοτροφών. Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα ε, στην παραγωγή σπόρων και στην έρευνα επίσης ε, και οφείλουμε να ελεξιτοποιήσουμε αυτό το έλλειμμα. Ζητούμε λοιπόν στην από την Εκτελεστική Επιτροπή να εξετάσει τον ενδεχόμενο ανάληψη τεχνικών μέτρων για να ε, το πετύχουμε. Ε, σας εξήγησα κάποια από τα πλεονεκτήματα αυτών των καλλιεργειών και εάν τελικά εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα που εισηγούμε εγώ στην έκθεσή μου, Εάν συμπεριληφθούν στη μελλοντική γεωργική πολιτική, νομίζω ότι θα έχουμε σημειώσει σοβαρή πρόοδο. Ε, στο παρελθόν έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα επανειλημμένα και θα το ξανασυζητήσουμε. Ε, μιλώ για τις ε, ζωικές πρωτεΐνες. Ε, οι ζωικές πρωτεΐνες πλέον έχουν αμεληταίο ρόλο στις ζωοτροφές από την κρίση των τρελών αγελάδων και ε, το λέω προσεκτικά γιατί κρεμούν ε, στην ουσία ακόμη πολλά ζητήματα. Κάποιες ε, ζωικές ουσίες, ουσίες ζωικής προέλευσης ε, ισχυρίζονται κάποιοι ότι πρέπει να ε, εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. Εγώ θεωρώ ότι γενική λύση δεν μπορούμε να δώσουμε και θα πρέπει η αρμόδια επιτροπή να δει κατά πόσο μπορούμε να επιτρέψουμε ζωικές πρωτεΐνες ε, μέσα στις ζωοτροφές. Έχω διάφορες συστάσεις, έχω συμπεριλάβει λοιπόν διάφορες συστάσεις μέσα στην έκθεσή μου. Είναι μεγάλο αυτό το κομμάτι της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ε, θα έλεγα ότι είναι η ε, ραχοκοκαλιά της γεωρικής ε, παραγωγής. Τα τελευταία χρόνια έχουμε εγκαταλείψει αυτή την παράδοση στην Ευρώπη. Δεν ήμασταν αρκετά προσεκτικοί και τώρα πλέον είναι κατεπήγον το ζήτημα, πρέπει γρήγορα να σημειωθεί η πρόοδος. Συζητήθηκε το θέμα στην Ολομέλεια, διαπιστώσαμε μεγάλε δυσκολίε ε, στον τομέα τη ε, κρεατοπαραγωγή ε, στην Ευρώπη και αναφέρθηκε ότι πρέπει να επιληθεί το ζήτημα των πρωτεϊνούχων. Νομίζω ότι μπορούμε να επεξέλθουμε σε αυτέ τι δυσκολίε αν ακολουθούν τα μέτρα που προτείνω μέσα στην έκθεσή μου. Έχουμε ήδη συζητήσει με του σκιώδει εισηγητέ και νομίζω ότι ακολουθούμε ε, το σωστό δρόμο. Ε, ε, έχουμε πολυάριθμες προτάσεις μέσα στην έκθεση και νομίζω ότι έτσι θα συνεισφέρουμε στην μεταρρύθμιση κοινή γεωργική πολιτική. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε. Μάρτιν, τώρα θα περάσουμε στη συζήτηση. Ο κύριο είναι ο πρώτο που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα εδώ δεν είναι μόνο τα πρωτεϊνούχα, αλλά ξεπερνάει κατά πολύ. Κατά πολύ. Τα πρωτεϊνούχα αποτελούν δείκτες, δείχνουν ότι υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα, μία διαμάχη. Δείχνουν ποιες είναι οι διαφορετικές θέσεις που τίθενται εδώ. Απ' τη μία οι ελεύθερες συναλλαγές και ζωοτροφών και τροφίμων που είναι τμήμα της παγκόσμιας αγοράς και από την άλλη μεριά το θέμα της τροφιμική μας αυταρκίας. Το κάθε κράτος μπορεί να διαλέξει μία από τις προτεραιότητές του. Τα πρωτεϊνούχα στην Ένωση προέρχονται από τη διεθνή αγορά και εν ονόματι των κανόνων της τελικά επηρεάζουμε και το περιβάλλον αλλά και καταστρέφουμε το 70% των καλλιεργειών μας εισάγοντας 80%. Καταστρέφουμε μάλλον το περιβάλλον στη Λατινική Αμερική. Τα πρωτεϊνούχα αυτά, τις πρωτεϊνούχες ζωοτροφές, τις εισάγουμε λοιπόν στην Ένωση από παντού και έτσι δεν καταστρέφουμε μόνο το περιβάλλον της αναπτυσσόμενης χώρας αλλά και το δικό μας περιβάλλον. Πώς χρησιμοποιούνται οι ζωοτροφές αυτές σε μερικές χώρες που διαθέτουν μεγάλα λιμάνια υπάρχουν μεγάλα πτηνοτροφία παραδείγματος χάρη και γι' αυτό ε, βιομηχανικού σχεδόν χαρακτήρα, πτηνοτροφία και εκεί κατευθύνονται τα πρωτεϊνούχα. Αυτό θέλουμε όμως. Αυτό εννοούμε βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλουμε δηλαδή η κοινωνία έτσι να δουλεύει. Όχι μάλλον. Πώς θα το λύσουμε. Κάτε με, η απάντηση είναι το ελεύθερο διεθνές εμπόριο να μπορέσει τελικά να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαγορεύει την λήψη προστατευτικών μέτρων για το περιβάλλον. Να βρούμε μια υγιή ισορροπία μεταξύ ελευθερίας και διακανονισμού για να αποτελέσει εκ νέου το κέντρο ο πολίτης στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας. Συνάδελφοι που πήγαν στην Ουγγαρία επισκέφθηκαν κτηνοτροφία και κτηνοτροφία και κτηνοτροφικές μονάδες και μας είπαν ότι υπάρχουν υγιείς επιχειρήσεις εφόσον μπορούν να εξάγουν ζωοτροφές Χρειάζεται δηλαδή εξισορρόπηση μεταξύ καλλιεργειών και κτηνοτροφίας, αγεωργίας και κτηνοτροφίας. Αυτό είναι το μόνο κριτήριο που μπορεί να μας εγγυηθεί τη βιωσιμότητα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την γεωργική αξιοπρέπεια και το περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τις μεθόδους μας και σας καλώ να το σκεφτούμε, να τη σκεφτούμε αυτή την αλλαγή. Ευχαριστούμε κυρία Μομπάη. Σας ευχαριστούμε και βεβαίως θα πρέπει τον κύριο Λάντερφέντερ να τον ευχαριστήσουμε μια που οργάνωσε αυτήν την αποστολή, την τόσο επιτυχή στην Ουγγαρία. Και θα συνεχίσουμε τώρα με την Μισελ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το συνάδελφό μας για αυτή την έκθεση. Γίνεται μια αρκετά ακριβής ανάλυση της κατάστασης για τις πρωτεονιούχες καλλιέργειες στην Ένωση και ανά τον κόσμο. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω επίσης ότι έχουν συναυθεί ε, παλαιότερα διεθνείς συμφωνίες στην εποχή της Ευρώπης των 15 ή και λιγότερων κρατών, ε, των 11, των 12, αν θυμάμαι καλά. Τότε η Κίνα δεν ήταν ο βασικός παίκτη τη ε, ε, παγκόσμια αγορά. Σήμερα έχει δημιουργηθεί μια νέα ισορροπία και άρα θα πρέπει να ε, επέλθει ένα νέο προβληματισμό και σημειώνται νέε τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Φυστού την προσοχή των μελών της Επιτροπής στα όσα γίνονται ανάμεσα στη Λατινική Αμερική και την Κίνα. Η Κίνα σήμερα γίνεται το πρώτο εισαγωγέα πρωτεϊνών με όρου παραγωγή πολύ λιγότερο απαιτητικού σε σχέση με άλλου. Άρα μελλοντικά θα εκτεθούμε σε αυτό τον κίνδυνο να μην είμαστε ο βασικότερος πελάτης, ο πιο ενδιαφέρον πελάτης αυτών των ε, προμηθευτών. Η ανακατανομή λοιπόν της τράπουλας στην Ευρώπη, η αύξηση της παραγωγικότητας στην κεντρική ε, Ευρώπη και η μεταρρύθμιση κοινή γεωργική πολιτική δημιουργούν μια πραγματική ευκαιρία την οποία θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε, δηλαδή αμυψίσπορα, ελάχιστη αμυψίσπορα στι ε, ε, καλλιέργειε τι ευρωπαϊκέ και να επιτρέψουμε νέε καλλιέργειε στην Ευρώπη, όχι έτσι απλά, αλλά με μακροπρόθεσμα μέτρα, γιατί ο τομέα των πρωτεϊνών πάσχει από διάφορα μειονέκτηματα. Πρώτον, η επιλογή των ποικιλιών ε, δεν γνώρισε την ίδια πρόοδο όπως η επιλογή των σιτήρων τα τελευταία 20-30 χρόνια. Επίσης, ε, η καταπολέμηση των παρασίτων, των συζανίων δεν έγινε ε, έρευνα, δεν υπάρχει λύση και άρα οι παραγωγείς απομακρύνονται από αυτές τις καλλιέργειες και δεν έχουν τη δυνατότητα ε, όρθα να ελέγξουν την κατάσταση. το health check, όπως είπε και ο εισηγητής στην παρουσίαση της έκθεσης, έδειξε ότι μπορούμε να έχουμε μια γρήγορη απάντηση για τους ε, παραγωγούς ε, δίνοντας μια, τονώνοντας και πάλι αυτήν την παραγωγή ε, θα έχουμε υποβάλει διάφορες τροπολογίες που συμπληρώνουν κάποια μέρο στοιχεία της έκθεσης αλλά ουσιαστικά συμφωνούμε με το περιεχόμενο δεν είναι βασικό το ζήτημα για την οικονομία, για τη γεωργία στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε Μισελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Χόισλινγκ για την έκθεση την οποία συνέταξε. Είναι πάρα πολύ αξιόλογη η έκθεση αυτή. Εν γέννη, συμφωνώ με αυτά που πρεσβεύει. Όμως, υπάρχουν τρία στοιχεία τα οποία θέλω να τα συμπληρώσω. Θέλω κάτι να πω για την ζωική πρωτεΐνη. Θα πρέπει να αναζητήσουμε κάποια λύση στην Ευρώπη σχετικά με αυτό το σημείο. Τι γίνεται. Με αυτά τα οποία τώρα αποτεφρώνονται ε, σαν, σαν υπολείμματα σφαγής, ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως κτηνοτροφή. Δηλαδή να χρησιμοποιούνται επιτυχώς αυτά τα υπόλοιπα, τα υπολείμματα, αυτά τα υλικά. Ας κάτσουμε να το μελετήσουμε, να δούμε τα αριθμητικά στοιχεία. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε πόσα τροποποιημένα κυκλοφορούν στην αγορά, γιατί και αυτό είναι μια μεταβλητή. Και κατόπιν αποκρισταλώσουμε μια θέση. Κάτι άλλο τώρα κάτι το οποίο με ενδιαφέρει πολύ. Πρόκειται για τις διμερείς συμφωνίες. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει και το ενδιαφέρον που θα προσδοκούσαμε για όλα αυτά. Λέμε τώρα για νέες συμφωνίες όταν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υπάρχουσες. Υπάρχει ας πούμε μια συμφωνία σημαντική με τον Καναδά. Να τις εξετάσουμε προσεκτικά. Διότι θα πρέπει το Κοινοβούλιο να έρθει σε επαφή με τον αρμόδιο επίτροπο. Θα πρέπει να έχουμε πιο δυναμική στάση και να προετοιμαστούμε για τα προβλήματα που θα προκύψουν στο μέλλον ο επόμενος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Και όντως υπάρχει πρόβλημα έλλειψης πρωτεινών στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν να κοφεύουμε και να θελοτυφλούμε. Αφού λοιπόν δεν πρέπει να γνωρίζουμε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να κάτσουμε και να προβλέψουμε τι ε, μελλοντικέ εξελίξει. Συμφωνώ με τα όσα λέει ο εισηγητή. Φυσικά και υπάρχει κάποιο κενό στην αγορά. Άρα θα πρέπει να επιφέρουμε κάποιες βελτιώσεις στις επιδόσεις μας ας πούμε για την ε, έρευνα. Θα πρέπει οι καλλιέργειες, οι πρωτενούχες να προαχθούν αλλά θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα της γραφειοκρατίας. και να δούμε πώς ε, δεν θα έχουμε γραφειοκρατία όσον αφορά τις ποσοστώσεις, όσον αφορά την καλλιεργούμενη επιφάνεια και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα τροποποιημένα και εν πάση δεν μπορούμε να επιβάλλουμε από τα πάνω όλες τις λύσεις. Συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Γέγκλε κατά τα άλλα για τα υποπροϊόντα κρέατος τα οποία προκύπτουν από τα σφαγεία και είναι σκάνδαλο το ότι αυτά που τρώνε άνθρωποι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για κτηνοτροφή ας πούμε χείρων. Αποτεφρώνονται πολλά από αυτά τα υλικά, τα παραπροϊόντα, τα υποπροϊόντα και τα υπόλοιπα στέλνονται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ας κάτσουμε και να το σκεφτούμε ορθολογικά. Μιλούμε πάντοτε για κάποια προϊόντα σφαγίων τα οποία είναι κατάλληλα για τον άνθρωπο. Ας είμαστε λογικοί και ας τα χρησιμοποιήσουμε και έτσι ας αρθεί αυτό το κενό που υπάρχει και φυσικά έχουμε αντιλήσει χρήσιμα συμπράσματα από την κρίση της εγκεφαλοπάθειας των βοηθών, όμως θα πρέπει να είμαστε λογικοί. Και εν τέλει θα να πω, συμφωνώντα και πάλι με την κυρία Γέγκλε, ότι θα πρέπει να κάτσουμε και να λάβουμε υπόψη το τι γίνεται στις διεθνείς αγορές, τι γίνεται με τα τροποποιημένα ε, και να κάτσουμε να εξηγήσουμε στον κόσμο τι ισχύει. Ίσως έχουμε εκτροπή των ε, εξαγωγών σε όμορες χώρες της Ένωσης, ε, στην Κίνα και τελικά να αναγκαστούμε το τελικό προϊόν να το εισαγάγουμε. Συμφωνούμε στις γενικές νομές της έκθεσης. Αλλά χρειάζεται να γίνουν κάποιες ε, μικροδιορθώσεις. Και πάλι σας ευχαριστώ και πάλι σας τονίζω το πόσο σημαντικές είναι οι ζωικές πρωτεΐνες οι οποίες είναι κατάλληλες προς ε, ανάλωση και κατανάλωση. Ας είμαστε λογικοί. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιάρ. Και τώρα ο κύριος Ταραμπέλα. Μα άκουσα τι είπαν οι συνάδελφοι κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ. Συμμερίζομαι τα συμπεράσματα και της έκθεσης την οποία χαιρετίζω στις συστάσεις της η έκθεση μιλάει για την τρομερή εξάρτησή μας από την Αμερικανική Ήπειρο και του Βορρά και του Νότου και ε, προβλέπει και μέτρα μείωσης της εξάρτησης αυτής μέτρα που ελπίζουμε να συμπεριληφθούν στη μελλοντική ΚΑΠ αλλά θα εγώ θέλω να επιμείνω σε ένα από αυτά ότι οι συμφωνίες του Blair House 91 με 93 είναι κάτι που πρέπει και αυτό να το αμφισβητήσουμε. Μας υπενθύμισε ο εισηγητή ότι υπογράφτηκαν σε διαφορετική εποχή, υπό διαφορετικές συνθήκες από τις σημερινές, σωστό αυτό, αλλά και σε διαφορετική συγκυρία. Από τότε συνήθισαν και άλλες διεθνείς συμφωνίες που είναι πιο σημαντικές από εκείνη, όπως το πρωτόκολλο του Κιώτου. Και εγώ θα έβλεπα θετικά, δεν ξέρω αν θα καταθέσω και μια σχετική τροπολογία, να είναι πιο δυνατή, πιο ισχυρή διατύπωση που να καταδικάζει τη συμφωνία αυτή του Blair House. Ο, βέβαια δεν είμαι νομικός, αλλά νομίζω ότι από άποψη διεθνούς δικαίου οι συμφωνίες αυτές του Blair House αντιφάσκουν με τις υπόλοιπες πια που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου κλπ. Όσα προβλέπει το Κιώτο τέλος πάντων. Και πέρυσι την Κοπεχάγη κάναμε μια προσπάθεια που ήταν η μια αποτυχία. Υπήρξε και η Κανκούν. Όλα αυτά ακυρώνουν τη συμφωνία του Blair House και ελπίζω να συμφωνήσουν οι συνάδελφοι και να εγκριθεί από κάποια πλειοψηφία στην Επιτροπή μας και ελπίζω και στο σύνολο του Κοινοβουλίου αυτή η αμφισβήτηση των συμφωνιών του Blair House. Να το πούμε ρητά. Γιατί νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε στο μέλλον να εφαρμόσουμε ελπίζω πραγματικά προγράμματα που να μειώνουν την εξάρτησή μας από τα πρωτεϊνούχα ή τα εισαγόμενα πρωτεϊνούχα. Σε ευχαριστούμε Μάρκο κύριος Ανιό. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Παρακολουθώ να μην ξεπεράσω το χρόνο. Τέσσερα στοιχεία θέλω να αφήσω Όπου η Ένωση έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα ως προς την προμήθεια πρωτεϊνών. Πρώτα απ' όλα οι από ψάρια. Για ξέρουμε ότι πάρα πολλά ψάρια χρειάζεται να τα απορρίπτουμε στη θάλασσα. Γιατί να μην τα χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα απορριπτόμενα ψάρια για ζωοτροφές. Εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Γιάρ επίσης και στα κόκαλα απορρίπτουμε πολλά. Γιατί τα κοτόπουλα να μην μπορούν να τρώνε κρέας. Γιατί. Χείριο μάλιστα και η χείρη κοτόπουλα. Εξάλλου από τα κόκαλα μπορούν να γίνουν και λιπάσματα. Όλα αυτά όμως εμείς τα πετάμε. Εδώ λοιπόν η απορρίθμιση είναι ουσιώδης. Τρίτος τρόπος που δυσκόλεψε τα πράγματα η Ένωση. Δέχτηκα μία αντιπροσωπεία Ρουμάνων Γεωργών, λοιπόν, που έφυγε ο Ρουμάνος αντιπρόεδρος, και μου είπαν ότι πριν πουν στην Ένωση καλλιεργούσαν γενετικώς τροποποιημένη σόγια. Αλλά τους είπαν ότι αν θέλουν να μπουν στην Ένωση πρέπει να σταματήσουν αυτή την καλλιέργεια. Τη σταμάτησαν λοιπόν, καλλιέργησαν φυσική σόγια και απέτυχαν. Και άλλες πρωτεΐνες χαμένες λοιπόν. Τέλος, δεν διευκολύναμε τίποτε και για τις εταιρείε που προσπαθούν να παραγάγουν ε, τα ζυζανιοκτώνα και παρασιτοκτώνα που θα χρησιμοποιηθούν για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων. Εδώ είναι πολύ αβάσιμα και αμφισβητήσιμα τα στοιχεία για την απαγόρευση. Αν όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη μας θα είχαμε επαρκή πρωτεϊνούχα, επαρκείς ποσότητες. Στο με... Και τώρα ο κύριος Ράιμερ και μετά ο Χωσέ Μποβέ. Σας ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση και θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Αναρωτιέμαι γιατί θεωρείται τόσο αρνητικό αυτό το έλλειμμα γιατί αυτόματα θεωρείται αρνητικό αυτό το έλλειμμα, μπορεί και να είναι θετικό, διότι έτσι μπορούν να υποφεληθούν άλλες χώρες, ε, εξάγοντας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κάλυψη αυτού του ελλείμματος. Έχουμε το έλλειμμα λοιπόν στις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, αλλά το ίδιο πρόβλημα έχουμε και με την παραγωγή γιατί η δική μας ε, κατανάλωση. Δεν είναι ο μόνος τομέας που παρουσιάζει έλλειμμα. Δηλαδή, η σόγια δεν είναι ε, μια πρωτεΐνη που κανονικά ε, χρησιμοποιείται αυτούς στις ζωοτροφές, χρησιμοποιείται το λάδι της σόγιας, ε, δηλαδή είναι ένα δευτερεύον προϊόν, ένα υποπροϊόν αυτό που χρησιμοποιείται στις ε, ζωοτροφές. Ε, δηλαδή καλλιεργούμε αυτή την πρωτεΐνη και ταυτόχρονα σημειώνεται και παραγωγή υποπροϊόντων. Λογικό είναι οι κάτοχοι των γεωργικών εκμεταλλεύσεων να μας πούνε ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι, ότι δεν λειτουργεί το σύστημα. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε πρόβλημα. Ε, επίσης ε, υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός και μείωση της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης. Υπάρχει λοιπόν ε, το ενδεχόμενο να έχουμε συγκριτικά πλέον εκτίματα λόγω του ελλείμματος αυτού. Μπορούμε σε ορισμένες χώρες ε, να καλλιεργήσουμε τέτοιους πρωτενούχους πόγους παραδείγματο χάρη, αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι σε όλες τις χώρες μπορούμε να καλύψουμε το έλλειμμα αυξάνοντας τις καλλιέργειες. Τα αμινοξέα επίσης για να περάσουμε στη σύνθεση των πρωτεΐνων έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, δηλαδή ορισμένε ζωοτροφές πρέπει να συμπεριλαμβάνουν υψηλό ποσοστό αμινοξέων. Ε, δεν σημαίνει ότι όλες οι πρωτεΐνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλες τις ζωοτροφές. Η σόγια ε, περιέχει πρωτεΐνες, ε, παραδείγματο χάρη, πρωτεΐνες ε, που ε, εύκολα μπορούν να χωνευτούν, να καταναλωθούν. Αλλά αυτό δεν ισχύει, παραδείγματο χάρη, για τον αρακά. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση και μιλάτε μέσα στην έκθεση για εξαναγκαστικό κανιβαλισμό. Δεν είναι μόνο αυτό. Ε, τι προσπαθούμε να κάνουμε, ε, ε, να βάλουμε τα, τους χείρους να τρώνε μόνο φυτικές πρωτεΐνες. Μα ο χείρος τρώει ό,τι βρίσκει στη φύση, αν δεν προσπαθήσουμε εμείς να τον ελέγξουμε. Υπάρχει Ε, μην ξεχνάτε επίσης ότι εισάγουμε ναι 70-80% των πρωτεϊνών, αλλά όσες προσπάθειες και να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε σημαντικά να μειώσουμε τις εισαγωγές μας. Τώρα, για τη σόγια και τα, τη γενετικά τροποποιημένη σόγια, ε, θα πρέπει νομίζω να συνεχιστεί ο διάλογος ε, αν δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε τις εισαγωγές, ε, ας τις πλαισιώσουμε, ας τις ρυθμίσουμε. Ε, γιατί δεν νομίζω ότι μπορούμε να αποφύγουμε τελείως ε, την γενετικά τροποποιημένη σόγια. Στην τελευταία μεταρρύθμιση όλα, όλοι θέλαμε την αποσύνδεση των ενισχύσεων. Ωραία. Άρα δεν θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την ε, παραγωγή με άμεσε ενισχύσει, γιατί αυτό αντιβαίνει στις διατάξεις ε, της προηγούμενης μεταρρύθμισης κοινή γεωργική πολιτική. σα ευχαριστούμε. Ο Ζωζέ Μποβέ και ο Λουίς Κάπουλο Σάντος ε, ακολουθούν. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή καθώς και όλους όσους συνεισέφεραν στην εξέταση του θέματος και τον συνάδελφο που ήταν στο γραφείο του Μισελ Μπαρνιέ όταν ήταν στη Γαλλία. Πολύ σημαντική η συμβολή του. Θέλω μόνο να κάνω δύο-τρία σχόλια. Η πρώτη για τον Blair House. Σήμερα πράγματι γίνεται νομική συζήτηση διεθνώς για τον Blair House. Μερικοί λένε ότι μας εμποδίζει και μας επιβάλλει μια, την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και άλλοι όπως και εγώ θεωρούν ότι το Blair House είναι από το 92 όπως είπε και ο Ταραμπέλας και ότι από τότε οι συμφωνίες του ΠΟΕ που οι ιδρυτικές συμφωνίες του ΠΟΕ συμπεριλαμβάνουν και το Blair House της ρήτρε του πιο ευνοουμένου κράτους. Μεταφέρθηκαν δηλαδή οι ρήτρε του Blair House ως προς την παραγωγή χόγιας σε όλες τις χώρες και μπαίνει η σόγια αφορολόγητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μηδέν φόρος. Αυτό ήταν το συμφέρον των ΗΠΑ. Η συμφωνία, η παλαιότερη των αρχών της δεκαετίας του 60, έγραφε ότι η Ευρώπη μπορεί να εξαγάγει δημητριακά, εμείς έλεγαν οι ΗΠΑ θα εξάγουμε πρωτεΐνες αλλά δεν θέλουμε να πληρώνουμε δασμούς. Και νομίζω ότι στους κανόνες του ΠΟΕ σήμερα δεν μας εμποδίζει πια το Blair House. Δεν μας επιβάλλει πράγματα όπως τον περιορισμό σε 5 εκατομμύρια εκτάρια την παραγωγή της χώγιας κλπ. Αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να το εξετάζουμε γιατί δεν έληξε η συζήτηση επ' αυτού. Υπάρχουν ακόμη διαφορές και διχογνωμίες και πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει ως προς το διεθνές δίκαιο. Δεύτερον, για το έλλειμμα. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι νομίζω ότι οι εισαγωγέ αυτές σόγιας που είναι από τους βασικότερους λόγους, αν όχι ο βασικότερος για το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών στα γεωργικά, είναι ακριβώς αυτός. Σήμερα η Ευρώπη έχει τέτοιο πρόβλημα λόγω των εισαγωγών σόγιας. Μπορούμε λοιπόν σήμερα να μειώσουμε την εξάρτηση αυτή, να μειώσουμε ίσως και να καταργήσουμε τελείως το έλλειμμα αυτό, αν μπορέσουμε να μετατρέψουμε ένα τμήμα των καλλιεργειών μας σε πρωτεϊνούχα. Το Γαλλικό Υπουργείο Γεωργίας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος έκαναν μελέτες που έδειχναν ότι με τη μετατροπή 7 μόνο της 100 των καλλιεργιών δημητριακών σε πρωτεϊνούχα θα μειωνόταν κατά 41% η εξάρτησή μας από αυτές τις αγωγές, σημαντικότατο ποσοστό. Και αν δεν περιοριστούμε στη σόγια αλλά και στο, στο σύνολο των πρωτεϊνούχων φυτών, το ίδιο ισχύει. Και αυτό ενδιαφέρει όλα μας τα ζώα και τα βοηδή και τους χείρους και τις κατσίκες και τα αρνιά. Επομένως, αφού ξέρουμε ότι είναι συγκεκριμένο το πρόβλημα πρέπει να το εξετάσουμε συγκεκριμένα και για το σύνολο των κτηνών μας, των μυρικαστικών, θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον οικονομικά να γίνει αυτή η μετατροπή. Άλλο που ήθελα να τονίσω είναι ότι σήμερα Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα στοιχεία ποιότητος, ε, κόκκινες ετικέτες κλπ. που να δείχνουν ότι οι πρωτεΐνες αυτές έχουν παραχθεί τοπικά και υγιεινά. Υπάρχει ακόμα, είναι και αυτό ένα εργαλείο για, που να δείχνει την ποιότητα της παραγωγής γιατί πολλοί αυτό ζητούν. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Και τρίτον, τα τροποποιημένα. Δεν θα ήθελα αυτή να είναι η βάση της συζήτησης. Μπορούμε να το δούμε, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα γενικά των ε, φυτικών πρωτεϊνών. Ακόμη και αν, παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες ε, αγροτικές επιχειρήσεις, Καργκίλ και άλλες, το έθεσαν, γιατί δημιούργησαν μονοπόλιο βέβαια, αυτό δεν ισχύει για την Νότια Αμερική και άρα δεν είναι το θέμα μας. Ας μην κάνουμε λάθος λοιπόν, ας μην θέσουμε αυτούς εκτός θέματος. Πρέπει να δούμε εάν οικονομικά ως προς την εναλλαγή των καλλιεργειών και το εμπορικό ισοζύγιο είναι πιο ενδιαφέρον ή όχι. Να παραγάγουμε μόνοι μας τις φυτικές πρωτεΐνες για να μειώσουμε την εξάρτησή μας ή όχι. Δεν είναι όμως το θέμα ποιο τύπος πρωτεϊνών τροποποιημένες γενετικώς ή όχι γιατί αυτό θα ήταν νομίζω λάθος συζήτηση. Ευχαριστώ. Πολύ καλά. Ευχαριστώ σας Ζεμποδέ και τώρα ο κύριος Λουίς Καπούλα Σάντος. Obrigado, eh, obrigado Presidente. Este é um debate muito importante. Ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συζήτηση και θυμηθείτε αυτά που συζητούσαμε την περασμένη εβδομάδα για τη μεταβλητότητα των τιμών των σιτηρών. Συγχαίρω τον εισηγητή γιατί θέτει ορθότατα το ζήτημα. Αλλά, συγγνώμη, δεν βλέπω συγκεκριμένες ε, λύσεις και θα έπρεπε ίσω, γιατί τι θα κάνουμε, θα τροποποιήσουμε τους διεθνείς κανόνες, ε, το είπαν και οι συνάδελφοι, θα είναι δυσχερέστατο αυτό. Ή θα δημιουργήσουμε όρους τόσο ώστε να αυξήσουμε τη δική μα εγχώρια παραγωγή. Μπορούμε να έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρία. αν ε, δείξουμε φαντασία με τη μεταρρύθμιση κοινή γεωρικής πολιτική και πραγματικά ευελπιστώ αυτή η έκθεση και οι τροπολογίε να σα εμπνεύσουν για να ακολουθήσουμε αυτή τη σωστή οδό στη μεταρρύθμιση. Τρίτο στοιχείο το θέμα των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών και των κρέαταλεύρων. Ε, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε αυτές τις συζητήσεις. Εγώ θα προτιμούσα να επικεντρωθούμε σε αυτά που είναι εφικτά ε, βάσει του νέου μοντέλου της κοινής γεωργικής πολιτικής για να αυξήσουμε τη δική μας παραγωγή. Δηλαδή, η παραγωγή γιατί δεν παράγουν, γιατί δεν είναι ανταγωνιστική. Ε, λοιπόν, τι να κάνουμε, να αλλάξουμε τα κίνητρα, να αλλάξουμε αλλάξουμε τους κανόνες για να γίνουν ανταγωνιστικοί. Αυτή είναι η πρόκληση στην οποία ε, καλούμεθα να αντεπεξέλθουμε και ελπίζω να μας βοηθήσει ο εισηγητής με την έκθεσή του, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έχει τόσες πολλές συγκεκριμένες προτάσεις μέσα αυτή η έκθεση. Πολύ σας ευχαριστούμε, Λουίς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Χόσλιν για την έκθεση που εξεπώνησε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογη. Αλλά Ίσως θα πρέπει να επιφέρουμε μία-δύο προσθήκες σε αυτήν για να την κάνουμε ακόμα καλύτερη και σε σχέση με αυτό το οποίο είπε ο Ράινερ, ίσως θα πρέπει να πούμε ότι η έλλειψη γίνεται όλο ένα και πιο έντονη και ε, φυσικά και στη Γερμανία έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε αμέσως να βρούμε τη λύση, θα πρέπει να ανεχθούμε την κατάσταση αυτή ε, και βέβαια μια που είναι τόσο μεγάλη η έλλειψη των πρωτεϊνών ίσως θα έπρεπε να την συμμαζέψουμε εάν κάνουμε αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι όπως η κυρία Γέγκλε και έτσι το έλλειμμα θα συρρυκνωθεί και θα είναι καλύτερα πράγματα για την Ευρώπη επίσης που χρηματιζόμαστε ε, όσον αφορά το, αυτό το οποίο αποφασίστηκε για την συμφωνία με τις ΗΠΑ διότι έτσι σε ορισμένε περιοχέ τη Ευρώπη υπάρχει ακόμα πιο έντονη έλλειψη, όπω α πούμε στην Βαβαρία. Εκεί πάρα πολλέ καλλιέργειε. Ε, έχουν υποστεί κάποιες καταστροφές, έχουμε προσπαθεί να χρησιμοποιήσουμε βιομάζα, αλλά εκτός από τη στήριξη ανά εκτάριο η τα υπόλοιπα μέτρα ε, υποστήριξης των καλλιεργειών τελικά δεν απέδωσαν. Είχαμε 10.000 τόνους παλιότερα και τώρα έχουμε κατέβει 2.800 τόνους και μιλούμε για 1.000 εκτάρια παλιότερα και τώρα που τώρα έχουν και αυτά πάρα πολύ μειωθεί. Άρα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ θα πρέπει να αλλάξουμε στάση και όσον αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί αν έχουμε 10 τόνους που μπορούν να παραχθούν όσον αφορά μια ποιοτική κτηνοτροφή. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει να έχουμε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις σε διάφορα σημεία της Ευρώπης. Και όπως προείπα Και όσον αφορά την κτηνοτροφία για βοηδή, έχουμε 10.000 τόνους ανεκτάριο και έχουμε αυτάρκεια και δεν χρειαζόμαστε εισαγωγέ για τις κτηνοτροφές των βοηδών. Επομένως, στην πράξη νομίζω ότι μπορούμε να σημειώσουμε κάποια πρόοδο και νομίζω θα πρέπει επίσης να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση γιατί έτσι θα είμαστε λιγότερο εξαρτημένοι από τις εισαγωγές. Τώρα για να γυρίσω στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε, νομίζω ότι εάν αρθεί αυτή η έλλειψη θα είναι κάτι πάρα πολύ ωφέλιμο. Ε. Πρόεδρος. Κύριε Αντιπρόεδρε, Πόλσον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω θα πρέπει να προβληματιστούμε σοβαρά και επανειλημμένα πριν σημειωθεί πρόοδος. Εγώ ήμουν εισηγήτρια για διάφορους κανονισμούς μεταξύ των ζωικά υποπροϊόντα, ε, για τη ρύθμιση των ε, κρεαταλεύρων και ηχθιαλεύρων. Και το έχω πει και πριν από 10 χρόνια το είπα έχουμε νέα επιστημονικά στοιχεία στη διάθεσή μας και αυτή τη στιγμή τολμούμε να πούμε ότι ήρθε η στιγμή να αναθεωρήσουμε τις αποφάσεις για τις ζωικές πρωτεΐνες. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η νομοθετική ρύθμιση του παρελθόντος έγινε σε πανικό. Θυμηθείτε τι γινόταν με τις διοξίνες, τα σκάνδαλα, ε, την αγορά τροφίμων στην Ευρώπη που, όπου επικρατούσε πανικός και χάος. Σήμερα λοιπόν έχουμε λύσει πολλά από αυτά τα προβλήματα και πολλά δεν ήταν και τόσο άσχημα αρνητικά όσο νομίζαμε. Θα πρέπει λοιπόν να το έχουμε αυτό κατά νου στις μελλοντικές συζητήσεις μας. Τα μυρικάστικα δεν πρέπει να τρέφονται με ε, κρεατάλευρα ούτε και με ηχθιάλευρα. Δεν πρέπει να τρέφονται με ζωικές πρωτεΐνες. Νομίζω όλοι θα συμφωνήσουν γι' αυτό. Οπότε όταν μιλάμε για καλλιέργεια πρωτεϊνών για ζωοτροφές, είναι σημαντικό να ξέρουμε τι ισχύει για τα κρεατάλβερα και τα Ε, γιατί όλος αυτός ο κλάδος εξαρτάται από τις πρωτεΐνες ε, υψηλής τρεπτική αξίας. Τώρα έχουμε το θέμα των χείρων και των ε, πουλερικών ε, γενικότερα. Εντάξει, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφύγουμε τον κανιβαλισμό. Δεν πρέπει να δίνουμε ε, στα ζώα να τρώνε ε, ζώα του ιδίου είδους ε, διατρέχουμε έτσι μεγάλους κινδύνους. Τα γουρούνια δεν τρώνε γουρούνια, εκτός αν πρόκειται για επίγουσα κατάσταση. Το ξέρουμε αυτό αλλά υπάρχει ένα σημείο που ακόμη δεν το έχουμε εξετάσει επαρκώς. Δηλαδή, εάν αφαιρέσουμε όλα τα υλικά κινδύνου ε, από τα σφάγια των βοηδών, και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ζώα που έχουν απλώς ε, πεθάνει αντί να βασιζόμαστε μόνο στα εγκεκριμένα σφάγια. Δεν είναι αυτό μια λύση. Κανείς δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Οι χείροι και τα πουλερικά δεν μπορούν πάντως να τρώνε πρωτεΐνες βοηδών. Αυτό το πράγμα είναι ουσιαστικό, είναι ένα ζήτημα ουσιαστικό και δεν έχει απαντηθεί με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι σαφές ότι οι ζωικές πρωτεΐνες που έχουμε δεν θα αντικαταστήσουν ολόκληρη την παραγωγή της σόγιας. Παρόλα αυτά είναι τόσο υψηλής θρεπτικής αξίας αυτή, αυτές οι πρωτεΐνες ε, που από περιβαλλοντικής άποψης πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το κόστος αυτών των υλικών. Άρα μήπως να εξετάσουμε κάποιες άλλες ε, λύσεις, δηλαδή να επανεξετάσουμε το ζήτημα πριν όλα ε, ανακατευθούν και γίνουν βιομάζα, αχταρμάς δηλαδή. Ευχαριστούμε την Αντιπρόεδρο Πάολσεν. Θυμάστε την περασμένη εβδομάδα η Επίτρο στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια της συζήτησης ε, του ψηφίσματος για το ζωοτεχνικά ζητήματα ε, υπευλήθη μια τροπολογία που εγκρίθηκε και που συνέβη με αυτά που μας λέει ο Αντιπρόεδρος Πάουλσον. Πάζω συμφωνώ μαζί της. Τώρα θα δώσω το λόγο στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Βάνσλεν. Βερσέλεν. Ναι, Βερσέλεν. Ζητώ συγγνώμη που παρέφερα το όνομά σα. Βερσέλεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και από την πλευρά της Κομισιόν καλωσορίζουμε τη σημαντική αυτή έκθεση για την έλλειψη πρωτεϊνόχων στην Ένωση. Γνωρίζετε, το είπε και ο εισηγητής, ότι πρόκειται για πρόβλημα που συζητιέται από τότε που πρωτοήρθα από το 78. Και πάντα λέγαμε τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση και τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι τώρα από τα μέτρα που λάβαμε δεν ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικά. Πάντως το θέμα ενδιαφέρει ακόμα η περίφημη συμφωνία του Blair House που ανέφερε και ο κύριος Μποβέ και άλλοι για αυτήν το 1992 είχαμε πει μόνο 5,4 εκατομμύρια εκτάρια να πρέπει να δεσμεύονται από τη συμφωνία αυτή. Αλλά από τότε άλλαξε τα πράγματα και η συμφωνία Blair House δεν εφαρμόζεται πια. Άρα, έχουμε βέβαια φτάσει σε παραγωγή 11 εκατομμύριων εκταρίων, πολύ πέρα του 5,4% που είχε αρχικά συμφωνηθεί. Και αν δούμε ποια ήταν η ανάπτυξη της παραγωγής πρωτεϊνούχων τα τελευταία τρία χρόνια, έχουμε ακόμη έλλειμμα, αλλά από 28,5% ανήλθαμε σε 35,2% των αναγκών μας. Άρα μειώσαμε λίγο την εξάρτηση χάρη στα βιοκάφουσιμα, λέει ο μιλητής. Όπως είχα πει λοιπόν, η έκθεση αυτή είναι πολύ επίκαιρη γιατί και εμείς πρόκειται να αρχίσουμε συζητήσεις για την πολιτική μας μετά το 2013 και η Κομισιόν θα κάνει τις κατευθυντήρες γραμμές της, θα διατυπώσει πολύ σύντομα. Ο συγκητής ήδη όμως αναφέρει κομμάτια της έκθεσης αυτής που ακόμη δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Δεν έχει καν εγκριθεί. Λέει, κάπου αναφέρει όμως την ημερομηνία 17 Νοεμβρίου πρέπει να τη διορθώσει να την κάνει 18 Νοεμβρίου γιατί τότε αποφασίσαμε ότι θα εγκριθεί. Α, ναι, βέβαια, βέβαια, λέει ο πρόεδρος. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για τα τελικά. Ορίστε Μάρτιν. Κοιτάξτε, Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που έκαναν προτάσεις και σχόλια. Βασικά θα ήθελα να τονίσω ότι, ότι λέγω, εδώ στην Επιτροπή μας πρέπει να δούμε τα βασικά στοιχεία, όχι τα δευτερεύοντα. Τα βασικά, τα κοινά σε όλα τα προγράμματα λένε ότι η κατάργηση της βοήθειας ή των επιχορηγήσεων δεν διευκόλυνε τίποτα. Εδώ μπορεί να διαφωνώ. Μακροχρόνια πρέπει να δούμε, μακροπρόθεσμα, αν αλλάζουν τα πράγματα ή όχι με τις επιχορηγήσεις. Μιλήσαμε για ζωικές πρωτεΐνες. Εγώ δεν το λέω στην έκθεσή μου αλλά είναι κάτι που πρέπει να το αναφέρουμε αργά ή γρήγορα. Συμφωνούμε όλοι. Ζητάω λοιπόν από την Κομισιόν το εξή. Επειδή υπήρξαν πολλά σκάνδαλα τελευταία που δείχνουν ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα και να υπάρξει κάποιος έλεγχος, ο οποίος όμως είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιβληθεί, Υπάρχει γι' αυτόν τον λόγο ο κίνδυνος να υπάρξουν και νέες καταχρήσεις αν δεν ελέγξουμε τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε ιδιαίτερα το θέμα των ζωικών αυτών πρωτεϊνών. Πολλές φορές εξάγουμε ζωοτροφές που δεν έχουν εγκριθεί και κατανάλωση στην Ευρώπη. όπως υπόλοιπα κοτοπούλων που εξάγουμε στην Αφρική. Αυτά βέβαια είναι προβλήματα πολυτελείας. Είναι ότι έχουμε πολλά υπόλοιπα τα οποία εξάγουμε στην Αφρική. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να γίνει ο έλεγχος. Υπάρχει το πρόβλημα του κανιβαλισμού που επιβάλλουμε στα ζώα και υπάρχει και η δυσκολία να τα δεχθούν όλα αυτά η κοινή γνώμη. Τώρα η γενετικώς τροποποιημένη σόγια. Την έκθεσή μου επίτηδες δεν αναφέρθηκα ρητά σε αυτό το θέμα. Δεν θέλω εδώ να κάνουμε συζήτηση που βασικά αφορά άλλο θέμα. Εγώ λέω απλώς το εξής. Το εξής. όσο περισσότερα πρωτεϊνούχα παραγάγουμε εμείς στην Ευρώπη τόσο μικρότερη θα είναι η εξάρτησή μας. Ορίστε λοιπόν η εναλλακτική λύση, ορίστε η λύση μάλλον. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει δοθεί άδεια για να είναι γενετικώς τροποποιημένη η σόγια. Στη Βραζιλία πολύ μεγάλο ποσοστό της σόγιας που καλλιεργείται και στην Αυστρία επίσης είναι γενετικώς τροποποιημένη. Και παρόλα αυτά υπάρχει η έλλειψη. Πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα. Διαφορετικά από αυτά που ισχύουν ήδη. Πολλοί ανέφεραν τη συμφωνία του Blair και μας λέει η Κομισιόν δεν ισχύει πια, δεν εφαρμόζεται. Αυτό με εκπλήσει κάπως. μας λέτε ότι έχει πάει στον σκουπιδότοπο της ιστορίας. Αν δεν εφαρμόζεται, αν δεν ισχύει πια αυτή η συμφωνία κύριε και κύριοι της Επιτροπής, τότε μπορούμε να τη διαγράψουμε τελείως. Πέστε το μας τότε όμως, ρητά. Αν το εμπορικό μας πρόβλημα, εμπορικό μας λέγω πρόβλημα, όπως η αφορολόγητη εισαγωγή σόγιας. Αποτελεί πρόβλημα και αυτό να το πούμε. Είναι λοιπόν λίγο αφηρημένα αυτά που μας λέει η Κομισιόν. Δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι ακριβώς η στάση της ως προς τον Blair House. Τι ισχύει, τι δεν ισχύει από εκείνη τη συμφωνία. Κυρία Ράιμερς τώρα. Πραγματικά καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχουν δύο λογικές, αλλά γενικά οι ελεύθερες συναλλαγές είναι κάτι που το δεχόμαστε, απλώς μπορεί να μας θέσει και ορισμένα ερωτήματα, απορίες, ανησυχίες. Γιατί το έλλειμμα μας 80% είναι τεράστιο στο ισοσύγιο πληρωμών μας. Τεράστιο. Θυμάμαι πολύ καλά το, τη συζήτηση που είχαμε οργανώσει εδώ στην Επιτροπή μας όπου είχαμε πει ότι η Ευρώπη βασικά δεν παράγει πια, δεν έχει αυτάρκεια σε σόγια αλλά ότι παράγει για την Κίνα. Τι θα γίνει λοιπόν στο μέλλον με αυτό το έλλειμμα στο ισοζύγιο με τη σόγια. Άκουσα και τον Αλβέρτο Ντες Στη Γερμανία δεν υπάρχει πρόβλημα μόνο με το ελαιόλαδο, είναι και το πρόβλημα της βανάνης. Αλβέρτε. Πρέπει λοιπόν να διαφοροποιηθούν οι καλλιέργειες για να μειωθεί το έλλειμμα. Και τα ελαιούχα είναι τμήμα των παραδοσιακών ευρωπαϊκών καλλιεργειών. Ενώ τώρα σιγά σιγά τα καταστρέφουμε και αυτά. Καταρχήν είναι πολιτιστικό οικονομικό πρόβλημα να χαθούν όλα αυτά, αλλά χάνουμε και γεωργικές ευκαιρίες. Είναι μεγάλα προβλήματα αυτά λοιπόν. Ένα είδος δηλαδή, μια ποικιλία αν θέλετε, να μην καλλιεργείται πλέον και να μην αναπτύσσονται νέες ποικιλίε, να μην γίνεται έρευνα. Υπάρχουν εδώ μεγάλες δυνατότητες και θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τέτοιου είδους καταστροφές ή απώλειες. Χαίρομαι πάντως ιδιαίτερα για όλα όσα είπαν οι συνάδελφοι που τα βρήκα πολύ επικοδομητικά. Εγώ δέχομαι <coughs> να διευρυνθεί το θέμα σε όλα όσα είπατε κι εσείς. Το σημαντικότερο από όλα βρίσκω ότι είναι στη μελλοντική ΚΑΠ να ληφθούν επίσης υπόψη όλα αυτά για τα πρωτεϊνούχα και από τη στιγμή που θα συμφωνήσουμε τότε τα υπόλοιπα θα λυθούν μόνα τους. Ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε επικοδομητικούς συμβιβασμούς. Γιατί μόνο με μια δυνατή έκθεση και ενιαία στάση θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Τουλάχιστον αυτό ελπίζω. Κάλιστα, Μάρτιν. Καλή τύχη. Και ως συνήθως θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε συμβιβασμούς όσο δυνατόν ευρύτερους. Περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το λεγόμενο 6. Η Ευρώπη ως πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο. Νέο πολιτικό πλαίσιο για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Ο τουρισμός κυρίες και κύριοι είναι πολύ σημαντική οικονομική δραστηριότητα ε, και για την απασχόληση. Η διαφοροποίηση της τουριστικής μας προσφοράς είναι κάτι το απόλυτα ζωτικό αν θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Και άρα ο αγροτικός τουρισμός επίσης πρέπει να παίξει το ρόλο που του ενδημόζει εισηγητής ο Αντιπρόεδρος Νικουλέσκου, στον οποίο δίνω αμέσως το λόγο για να μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής του. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει ο κύριος Νικουλέσκου. Ξεκινούμε με κάποιε λεπτομέρειε και διευκρινήσει. Ε, με την συνήθεια τη Λισαβόνα έχουμε κάποιε τέτοιε αρμοδιότητε για ζητήματα τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακριβώ ε, και με αφορμή αυτέ τι ε, νέε αρμοδιότητε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει μαζί με τα κράτη-μέλη και μαζί με τους εμπλεκόμενους στην πολιτική του τουρισμού να δημιουργήσει ένα καινούργιο πλαίσιο για μια πολιτική τουρισμού και σύμφωνα με την ε, Επιτροπή θα πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να βοηθήσουμε το να υπάρχει ένας ε, αηφόρος, βιώσιμος τουρισμός, ε, ποιοτικό, θα πρέπει να την κάνουμε πιο διαρκή, πιο, πιο, πιο στέρεα την καλή εικόνα της Ευρώπης και έτσι να υπάρχει και κάποιο χρηματοοικονομικό μέσο και, και πρικοδότηση αυτής της πολιτικής. Όμως έτσι θα πρέπει να υπάρχει επίσης και κάποια ποικιλία, θα πρέπει να υπάρχει επαγγελματισμό από σε αυτών που εργάζονται στον τουρισμό, θα πρέπει να πιάσουν τόπο οι γνώσεις μας, ε, οι κοινωνικο-οικονομικές για τον τουρισμό και θα πρέπει μέσα αυτός ο βιώσιμος τουρισμός να στηρίζεται στην πρόθεση της εικόνας της Ευρώπης και έτσι να προβάλλεται περισσότερο η Ήπειρός μας. Οπότε η Επιτροπή εδώ προτείνει μια σειρά δράσεων και προτείνει επίσης τη δημιουργία ενός αυθεντικά ευρωπαϊκού πλαισίου για να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τις δυνατότητές μας και, και τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Επίσης μιλούμε για πάρα πολλά προγράμματα τα οποία σήμερα τρέχουν ε, στα πλαίσια της ΚΑΠ. Μετά το 2013 όμως δεν υπάρχει κανένα είδους συγκεκριμένη δέσμευση. Όμως υπάρχουν διάφορες δυνατότητες ώστε να βοηθήσουμε τον τουρισμό ε, και έτσι να βοηθήσει αυτή η πολιτική στην υλοποίηση των ε, προτεραιοτήτων μας. Και θεωρούμε ότι χρειάζεται μια έκθεση πάνω σε αυτό το θέμα. και να συνεχίσει η Ευρώπη να έχει τον πρωτενιστικό ρόλο το οποίο έχει και θα πρέπει και εμεί πρώτη-πρώτη να περνούμε τι διακοπέ μα στην ύπεθρο, ε, στην εξοχή, σε μικρά αγροκτήματα ε, και στι μικρέ πανσιόν ε, γιατί ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι ο αγροτουρισμός. Ο, μιλούμε τώρα για 500.000 καταλήμματα που υπάρχουν. Ε, έχουμε 6 εκατομμύρια κλίνες και μιλούμε για 10-15% της αύξησης σε αυτές τις ε, δυνατότητες. Πάντως η αύξηση τουρισμού ε, κινείται στο 4 με 5%. Άρα ο κλάδος αυτός αξίζει τη προσοχή μας. Και επίσης να βελτιωθούν τα πράγματα στην Ήπεθρο. Και έτσι να αποφύγουμε την απερίμωση της Ήπεθρου. Γιατί και η πολιτική ταυτότητα δεν είναι άσχετη με την υπόθεση αυτή. Άρα, να αναπτυχθεί ο αγροτουρισμός. Και θα πρέπει να διατυπώσουμε προς την Επιτροπή της προτάσεις μας. Να επιμείνουμε στο ότι θα πρέπει οι δράσεις της Φέντεραρ να στηριχτούν και χρειάζεται επίσης και χρηματοοικονομική στήριξη, χρειάζονται κάποια μέτρα για να, <clears throat> να προσθεθεί η ΚΑΠ και κάποιες άλλες δράσεις ούτως ώστε ε, αυτός ο αγροτουρισμός να στηριχτεί και έτσι να αναπτυχθεί η Ήπεθρος, να συντηρηθεί, να διασωθεί η κληρονομιά μας και με την πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρησιμοποιηθούν και οι καινούργιες τεχνολογίες. Επίσης με αυτόν τον τρόπο πρόκειται η να έχει προσβασιμότητα στις νέες τεχνολογίες, συγκεκριμένα και στο ίντερνετ και ασύρματη πρόσβαση αλλά, από την άλλη μεριά, εδώ έχουμε και θέμα γεωργικών προϊόντων. Αλλά αυτά τα ξέρετε. Θα πρέπει επίσης η πρωτοβουλία καλύψω και μετά το 2012 να συνεχίσει να τρέχει. Πρόκειται για κάποιες ε, αλλαγές και πέραν της καθεαυτού τουριστικής περίοδου. Καλύπτει και τους ηλικιωμένους και τους νέους αλλά και τους αναπήρους. Έτσι επομένως θα βοηθήσουμε και τον τουρισμό στην Ήπεθρο και τον αγροτουρισμό. Θα αναπτυχθεί έτσι η Ήπεθρος, οι αντίστοιχε ζώνες, αλλά επίσης και οι παραμεθόριες περιοχές. Είναι συγκεκριμένοι αυτοί η χώρα πεπερασμένη. και πιστεύω ότι οι τροπολογίες σας θα βελτιώσουν το κείμενό μου. Και τώρα να το συζητήσουμε, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Λουίς Καπούλα Σάντος θα λάβει τον λόγο. Και θα είναι ο κύριο Μπρέκοβιτς, ο Αντιπρόεδρος. Θα ήθελα να ε, επιχαίρω μάλλον για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί ο τομέας του τουρισμού δημιουργεί περισσότερη απασχόληση από πάρα πολλούς και ε, ε, στη, κυρίως σε αγροτικές περιοχές, στην Ήπεθρο. Οπότε μπορούμε να τονίσουμε αυτήν την πτυχή του αγροτουρισμού ε, στο μέτρο του δυνατού και ελπίζω με την παρέμβασή μου να συμβάλλω κι εγώ. Θα ήθελα να πω στον εισηγητή μας ε, το εξή. Θα, νομίζω θα ήταν καλό η Επιτροπή Γεωργίας ε, να προτείνει, όπως εξάλλου αναφέρεται μέσα στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχουν οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες. Λοιπόν, καλό θα ήταν να είχαμε τουριστικές πολιτιστικές περιφέρειες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να εστιάζουμε σε άλλες περιοχές, όχι μόνο σε μία πόλη. Και έτσι θα τονίσουμε την ε, διάσταση αυτή του αγροτουρισμού. Επίσης ε, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ρυθμός της φύσης, γιατί ο αγροτουρισμός μας επιτρέπει να παρουσιάζουμε διαφοροποιημένα προϊόντα Δηλαδή ε, είναι εποχιακό φαινόμενο τα προϊόντα σε ορισμένο βαθμό. Υπάρχουν οι διακοπές ε, το καλοκαίρι και πάμε στην παραλία. Μην ξεχνάτε όμως ότι υπάρχουν οι συγκομιδές. Ε, υπάρχουν και άλλες εποχές του χρόνου όπου υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον και μπορούμε να προσεγγίσουμε νέους πελάτες σε περιοχές της υπαίθρου. Ε, και νομίζω ότι αυτό θα καλύψει και άλλες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, το αναφέρατε κι εσείς, ε, που είναι ολοένα και πιο πολυάριθμοι και έχουν και υψηλή αγοραστική δύναμη. Ε, δηλαδή, ο προσανατολισμό μα αυτό θα είναι να καλύπτουμε τέτοιε πληθυσμιακέ ομάδε αλλά και τι αναπτυσσόμενε χώρε. Δηλαδή, νέε ομάδε που έχουν αγοραστική δύναμη. Ε, νέε πληθυσμιακέ ομάδε νέων αναδυόμενων οικονομιών. Αυτό μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη του τουρισμού. Ε, και μην ξεχνάμε, δεν υπάρχει μόνο ο πολιτισμό, δεν υπάρχουν μόνο τα μνημεία. Πρέπει να γνωρίζουμε τι ρίζε ε, του πολιτισμού όλα καιρού και φυσικά πρέπει να γνωρίζουμε την παραδόσεις της υπαίθρου μεταξύ άλλων. Σας ευχαριστούμε, Λουίς, η Αντιπρόεδρος Πάουλσεν τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ μένω σε μια εξαιρετικά αεροκατοικημένη κοινότητα ε, που είναι με λίγο μεγαλύτερη από το Χέτιγκομ στο Λουξεμβούργο. 10.000 πληθυσμό έχει, έχουμε το, ε, τουρισμό λόγω του σκι ε, και έχουμε 65.000 κλίνες ε, στα ξενοδοχεία μας. Αλλά πρόκειται για χειμερινό τουρισμό. Σε άρεο κατοικημένες περιοχές της Υπέθρου λοιπόν αποδεικνύεται ότι μια τέτοια τουριστική δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη, σε θέσεις απασχόλησης ε, προστατεύοντας ε, την γεωργία και προγράμοντας την δασοκομεία. Δηλαδή, μπορούμε να προωθήσουμε τον αγροτορισμό χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτές τις εκτάσεις. Ε, είναι δυνατός ο τουρισμός και στα παράλια και στα βουνά. Ε, υπάρχει η δυνατότητα έτσι να επιδιώξουμε κοινού στόχου ανεξάρτητα από την περιοχή. Έχουμε πολιτιστικέ πρωτεύουσε, έχουμε τα μνημεία μα, έχουμε τι εκθέσει τέχνη. Όλα αυτά ε, έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την πολιτική μας κληρονομιά, αλλά βρίσκονται στις πόλεις. Αλλά συγγνώμη, 55% και παραπάνω του ευρωπαϊκού πληθυσμού σήμερα ε, μένουν σε πυκνοκατοικημένες αστικές ε, περιοχές. Ε, και όσο πιο πυκνοκατοικημένες είναι οι αστικές περιοχές, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι ανάγκες που δημιουργούνται για να νιώσουμε και λίγο τη φύση, την ησυχία, τη γαλή ειρήνη, την ηρεμία της ε, φύσης ε, ε, για να μπορέσουν να αναπτυχθεί και η ίδια η φύση και εμείς. Οπότε είναι σημαντικό να προαγάγουμε τον αγροτουρισμό, αλλά τονίζω σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα. Παραδείγματο χάρη, η γεωργία μικρή κλίμακα, η παραγωγή, η βιοτεχνική παραγωγή τροφίμων. Όλα αυτά μπορούν να προωθηθούν για να επιβιώσει η ύπεθρος, ε, κυρίως η εξόχως απομακρυσμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. E Ευχαριστούμε κυρία Πάουλσεν, Ντόρφμαν και μετά Ανιό. Ευχαριστώ πρόεδρε. η τουριστική αυτή πολιτική είναι ακόμα στην αρχή της. Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει νέες δικαιοδοσίες που τώρα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε. Τι είναι το πιο ενδιαφέρον λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε ενωσιακώς και τι δεν θα έπρεπε. Υπάρχουν πράγματα που έχουν συζητηθεί που δεν έχουν όμως μεγάλο ενδιαφέρον. Ο τουρισμός είναι θέμα περιφερειακό, τοπικό. Υπάρχει ο αγροτουρισμός, υπάρχει ο οροτουρισμός, υπάρχουν πολλές δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. Για κοινέ προτάσεις νομίζω ότι αυτές πρέπει να τις πάρουν οι παράγοντες του ιδιωτικού τομέα. Εκείνοι μπορούν να δώσουν μια νέα ορμή στις δραστηριότητες τους. Ας πούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία. Ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να μπούμε εμείς σε αυτά τα θέματα. Η αγορά θα δείξει ποια είναι η σχέση προσφοράς και ζήτησης και σε αυτά τα θέματα. Εγώ είμαι από περιφέρεια όπου έχουμε 50.000 κατοίκους και 28.000 κλίνας ή μονάδες, ε, κυρίως αγροτικές κλίνες. Και 2.000 άνθρωποι ασχολούνται με αυτό τον αγροτουρισμό. Με δύο τρόπους μπορούμε να δούμε το θέμα. Πρώτον, η γεωργία αφορά και τον τουρισμό, γιατί αν δεν υπάρχει ένα ωραίο τοπίο περιποιημένο στα βουνά, μιλάω για τον ορεινό τουρισμό, ε, δεν θα έρθουν οι τουρίστες. Η γεωργία λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την διατήρηση για να το πω έτσι του περιβάλλοντος για να είναι πιο ελκυστικό και η προσφορά αυτή των γεωργών των αγροτών και αγροτισών είναι κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και για τον τουρισμό. Το κοινό λοιπόν αυτό αγαθό είναι σημαντικό. Δεύτερον, η προσφορά κάθε καθεαυτήν. Αν οι αγρότες και οι αγρότησες συμβάλλουν στον τουρισμό ή μάλλον εφόσον συμβάλλουν, τότε πρέπει να έχουν και κάποιο όφελος από αυτό και είπε ο εισηγητής όλα όσα θα έπρεπε να γίνουν. Ο αγροτουρισμός πρέπει να βελτιωθεί, να αναπτυχθεί ίσως με κάποιες επιχορηγήσεις από το δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ γιατί η αγορά αυτή αναπτύσσεται, αναπτύσσεται. Πώς θα μπορούσαμε να τη βοηθήσουμε σε ορισμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες είναι γνωστό ότι μπορεί να υπάρξουν τεράστια ωφέλη. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος Ντόρφμαν. Θα μιλήσω και εγώ αργότερα, ο κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μπορεί να σας φανώ κοινικός, αλλά εμείς στη Μεγάλη Βρετανία κάποτε είχαμε πολύ ωραίο τοπίο. Έρχονταν τουρίστες να απολαύσουν το χόρτο μας και τον καιρό μας, ενώ τώρα, τώρα τι βλέπουν. Όλο τουρμπίνες. Τουρμπίνες και τώρα δεν έρχονται οι τουρίστες παρά για να δουν πόσα ψόφια πουλιά μπορούν να μετρήσουν κάτω από τις τουρμπίνες. Και εκτός από τις τουρμπίνες τώρα έχουμε και τους ηλιακούς συσσωρευτάς. Stop Επομένως, όλο και περισσότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που καταστρέφουν το τοπίο. Τι τουρισμό να αναπτύξουμε εκεί. Ωραία, έληξε η συζήτηση. Τώρα η Κομισιόν, η κυρία Χαλούνας. Ή Χαλούας μήπως, άμεση, συγχωρείτε, Χαλούας. Όχι, όχι, καλά το είπατε, Χαλούνας, Χαλούνας. Ευχαριστώ πολύ. Διότι πήρατε την απόφαση να μιλήσετε κι εσείς, να πείτε κι εσείς το λογάκι σας για αυτή την ε, ανακοίνωσή μας για τον τουρισμό και άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου θα γνωμοδοτήσουν επί του τουρισμού. Όπως είπε ο κύριος Λουπέσκου, λέει η ομιλήτρια, η ανακοίνωσή μας συνδέεται πολύ με τη συνθήκη της Λισαβόνας. συνθήκη της Λισαβόνας η οποία για πρώτη φορά αναγνωρίζει ενωσιακή δικαιοδοσία για στήριξη των κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού και της περιηγήσεως. Δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα, αυτό όλοι το γνωρίζουν και άρα οι δράσεις που προτείνουμε είναι απλώς στηρικτικές και συμπληρωματικές. Πέρα από τη συνθήκη της Λισαβόνας, η ανακοίνωσή μας στοχεύει να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας στρατηγική, αναπτυξιακής στρατηγικής 2020 στην οποία ο τουρισμός θα έχει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα διότι η ανταγωνιστικότητα είναι σημαντικό τμήμα αυτής της ανακοίνωσης και συνδέεται φυσικά και με την ποιότητα και τη βιωσιμότητα. Όπως τονίστηκε ήδη, τέσσερα, τέσσερις βασικοί πυλώνες έχουν αναφερθεί. Ανταγωνιστικότητα, βιωσιμότητα και ποιότητα, καθώς και ευθύνη, ευπευθυνότητα των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και την ορατότητα της Ευρώπης και των προορισμών της, όχι μόνο μέσω της προώθησης κοινών ποιοτικών ετικετών, αλλά και βοηθώντας άμεσα τα κράτη-μέλη και τους τουριστικούς τους οργανισμούς να καταλάβουν καλύτερα τις διαφορές μεταξύ αγορών και που θα έχουν τη δυνατότητα έτσι να προωθούν καλύτερα τους προορισμούς τους. Η τέταρτη προτεραιότητα είναι καλύτερος συντονισμός και καλύτερη συνεργασία σε ολόκληρη την Ένωση διότι ο τουρισμός είναι οριζόντιο πρόβλημα θέμα και ό,τι αποφάσεις ληφθούν στον τομέα της γεωργίας μπορεί να έχουν επιπτώσεις επί του τουρισμού ή επί του περιβάλλοντος και οι νομοθετήματα επίσης μπορεί να έχουν τέτοιες επιπτώσεις και άλλα. Για τον αγροτουρισμό τώρα δεν λέμε πολλά στην ανακοίνωσή μας διότι είχαμε τον περιορισμό του μεγέθους της ανακοίνωσης, γι' αυτό παραμείναμε τόσο ασαφείς. Κάναμε, είπαμε ορισμένα πράγματα, αλλά που θα αναπτυχθούν αργότερα κατά την εφαρμογή. Γι' αυτό είπαμε ότι θα υπάρξει και ένα δεύτερο περαιτέρω έγγραφο που θα συζητηθεί πρώτα την επόμενη εβδομάδα όχι αυτή την εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα στις 18 και 19 Νοεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Τουριστικό Βήμα με τα κράτη-μέλη και εκπροσώπους του τομέα τουριστικών οργανώσεων πανενωσιακός καθώς και με μερικούς βουλευτάς από διάφορες επιτροπές. Αυτή η ανακοίνωση, το πρώτο της τουλάχιστον σχέδιο, απλώς λέει γενικά πώς θα θέλαμε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τους εκπροσώπους του τομέα να εφαρμόσουμε τις προτινόμενες δράσεις. Χρειάζεται ακόμα βέβαια κάποια απλοποίησή τους διότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Θα ήθελα να, ευχαρισ... να σας ευχαριστήσω που αναφέρατε την πρωτοβουλία της Καλυψούς που είναι ένα πρώτο πρόγραμμα που ενέκρινε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που τώρα από το 2011 α, έφτασε στον τρίτο και τελευταίο χρόνο του και που έχει στόχο να βοηθήσει τον, την τουριστική βιομηχανία και τα κράτη-μέλη να ξεπεράσουν το πρόβλημα της εποχιακότητος ή τουλάχιστον να προσπαθήσουν να βρουν κάποια λύση για το πρόβλημα αυτό. Ο αγροτουρισμός πράγματι είναι πολύ σημαντική πτυχή του γενικότερου τουριστικού θέματος για τη διαφοροποίηση των τουριστικών μας δραστηριοτήτων. Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και στις μελλοντικές μας προτάσεις ελπίζουμε να μας βοηθήσουν, βασιζόμαστε στη βοήθειά τους ώστε να υπάρξει μια συνδυασμένη προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Α, ωραία. Ευχαριστώ την Κομισιόν. Τώρα ο Αντιπρόεδρος Νικουλέσκου για τις final remarks που λέμε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις απόψεις τους και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας διαβεβαιώ ότι σημείωσα όλες τις παρατηρήσεις σας και θα τις λάβω υπόψη κατά την σύνταξη της τελικής έκθεσης. Θα λάβω υπόψη δε και τις τροπολογίες. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τον συνάδελφο Χόφμαν και τις αρμοδιότητες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του τουρισμού, αληθεύει ότι υπάρχει τέτοια αρμοδιότητα. Εγώ νομίζω ότι στην Επιτροπή Γεωργίας συζητούμε για το δυναμικό που έχει ο αγροτουρισμός για την ανάπτυξη της οικονομίας της Υπέθρου και γενικότερα για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν γίνει σοβαρές επενδύσεις, υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά μέσα, τα διαρθρωτικά ταμεία που χρηματοδοτούν δράσεις για να προαγάγουν τον αγροτουρισμό. Δεν πρόκειται λοιπόν για καινοτομία. Ελπίζω ότι θα συνεχιστούν αυτά τα προγράμματα και σας ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ανοιχτό πνεύμα που δείχνει. Χάρη στις ενημερωτικές εκστρατείες και τα προγράμματα μπορούμε να βελτιώσουμε τις υποδομές. Ο αγροτουρισμός είναι ε, μία εναλλακτική λύση σε σχέση με άλλα είδη τουρισμού και μπορεί να ενδιαφέρει και τους Ευρωπαίους τουρίστες και τους τουρίστες τρίτων χωρών. Για να είναι βιώσιμη όμως αυτή η εναλλακτική λύση, πρέπει να γίνει πιο ελκυστική. Πιστεύω ότι είναι ευπρόσδεκτη αυτή η πρότασή σας, κυρίως για την προστασία της ε, υπαίθρου και θα λάβω υπόψη τις παρατηρήσεις σας. Ε, ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο Νικολέσκο. Θεωρώ ότι λίγη η συνεδρίαση. Αν σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει την 5η στις 18 στις 2, 2, 2 μετά μεσημβρίας ε, παρουσία του Επιτρόπου Τσιόλος στην αίθουσα 4Q2 αν δεν υπάρχει επαρκή θέση, θα υπάρχει πέρα από την 4Q1 και μία άλλη αίθουσα για τους ακρατες 4 4Q2 συγκεκριμένα. Θα παρουσιάσει ο Επίτροπος την ανακοίνωση για τη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική στις 2 το μεσημέρι την Πέμπτη. η ναι. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για την έκθεση Hoesling για τις πρωτεΐνες έχει τεθεί για την 29η Νοεμβρίου μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Αυτή είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες για την έκθεση Hoesling για το έλλειμμα πρωτεϊνών. 29 Νοεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Λουίς. Ε, συγγνώμη, στο, υπό τα διάφορα, στο σημείο 7, δεν είμαστε στο 7 τώρα, στα διάφορα, ωραία. Θέλω να θέσω ένα ζήτημα. Ε, να σας μιλήσω για τη συνάντηση με τον Επίτροπο Τσιόλος για την παρουσίαση της ανακοίνωσης για την κοινή γεωργική πολιτική. Διάφοροι βουλευτές μου είπαν πως ε, οργανώσεις γεωργών των χωρών τους ε, έκαναν κινήσεις, ε, έλαβαν προσκλήσεις ε, για να παραστούν στην παρουσίαση και δεν υπάρχουν πλέον θέσεις ούτε σε αυτή τη δεύτερη αίθουσα, μήπως χρειάζεται και τρίτη. Δεν θα υπάρχει αναμετάδοση με βίντεο, θα παρακολουθούν μόνο ηχητικά. Ωραία. Και εγώ ήθελα να προτείνω το εξή. Γιατί δεν πάμε στο ημικύκλιο. Ε, καλό θα ήταν η Επιτροπή Γεωργία ε, που ενδιαφέρεται φυσικά για την ανακοίνωση, καλό θα ήταν λοιπόν να φροντίσει ώστε η κοινωνία των πολιτών να μπορέσει να παραστεί ε, στην παρουσίαση της ανακοίνωσης. Θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την πρόταση, γιατί είναι νομίζω η μεγαλύτερη αίθουσα που διαθέτουμε. Εξαιρετική η ιδέα σας, Λουίς Κάπουλα. Σαντός ε, να διεξαχθεί συνεδρίαση στο ημικύκλο. να σας πω ότι την πρώτη απόπειρα την είχε κάνει η γραμματεία ήδη όταν μας το θέσατε το ζήτημα πρώτη φορά και προς το παρόν ε, λάβαμε, ε, έχουμε λάβει αρνητική απάντηση. Αν συμφωνείτε όλοι, ας επανέλθουμε, ας προσπαθήσουμε να πιέσουμε, γιατί έτσι θα γίνει η συζήτηση στο ε, ημικύκλιο και σίγουρα θα υπάρξει και μεγαλύτερη προσέλευση και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ε, τώρα, ο κύριος Άλβαρες ε, πάλι υπό τα διάφορα. Ναι, ήθελα απλώς να υποστηρίξω αυτή την πρόταση. 16 γεωργικές οργανώσεις από τη δική μου περιοχή θα παραστούν στην παρουσίαση. Πολύ καλό θα ήταν να μην υπάρξουν δυσκολίες, να μπορέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να παραστούν στην ίδια την αίθουσα στην παρουσίαση ε, της ανακοίνωσης. Σας ευχαριστούμε κυρία Άλβες λέει ο Πρόεδρος. Τώρα στρέφομαι προς όλες τις πολιτικές ομάδες. Αν έχετε κάποιες ενδείξεις σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών, των προσκεκλημένων, δώστε μας τα στοιχεία γιατί έτσι θα ε, στοιχειοδητήσουμε και καλύτερα την, ε, το αίτημα που θα υποβάλει εκ νέου η Γενική Γραμματεία. Ε, θα διακόψουμε δύο λεπτά, έτσι, αν συμφωνούν και οι συντονιστές και αμέσως μετά θα αρχίσουμε την συνεδρία των συντονιστών. Σας ευχαριστούμε. Λίγη συνεδρίαση.